τα μέλη Μάρτο Καπάτο, Κουμπίτσκα, Τόμας Μακτάνο και Χέλγκα Τριούπελ κατέθεσαν την ε, γραπτή δήλωση 26 του 2008 για την ε, εκπομπή του σταθμού TDTV στην ε, Κίνα κάτι το οποίο θα διαβιβαστεί σε αυτούς που απευθύνει σύμφωνα με το άρθρο 106 του κανονισμού και θα δημοσιευτεί στην συνεδρίαση του Φεβρουαρίου 2009. Τον λόγο σχετικά και ο κύριος Καπάτο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ε, θέλω να ευχαριστήσω εξ ονόματος όσων ε, ξεκίνησε την ε, συμβιβαστική αυτή λύση τους υπόλοιπους 440 βουλευτές που συνυπέγραψαν το κείμενο. Εμείς ζητάμε από την Utah να ξαναρχίσει τις εκπομπές της MTT TV στην Κίνα. Η ελευθερία της γνώσης είναι βασικό δικαίωμα του ανθρώπου. Το Κοινοβούριο δείχνει όπως ε, με το βραβείο Ζαχάροφ ή με την πρόσκληση στο Δαλάη Λάμα ότι όταν μιλάμε για τα δικαιώματα του ανθρώπου τα κάνουμε για να υποστηρίξουμε τον λαό, την ελευθερία του λαού της Κίνας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ακολουθεί τώρα η ψηφοφορία σήμερα με απλοποιημένη διαδικασία για την έκθεση της κυρίας Ματιέ για το Μουσουλμικό Έλεγχο των Κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αφγανιστάν. Ψηφίζουμε με ονομαστική ψηφοφορία, έναρξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Ναι, καθίστε παρακαλώ στις θέσεις σας.